παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Πρώτο θέμα είναι η κάταρτη τη ε, Κρυμαία. Ε, συνάδελφοι, έχουμε μείνει πίσω. Δεν θα δεχτώ μπλε κάρτε, σα ενημερώνω και ενδεχομένω να αναγκαστώ να μειώσω και τη διαδικασία Catch the Eye. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο στα πλαίσια του Catch the Eye σε κάποιου συναδέλφου, δεν το εγγυώμαι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση για του τατάρου τη Κρυμαία και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ροπέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα συζητούμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Τατάρους της Κρυμαίας. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτή τη μοναδική εθνοτική ομάδα. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι όλοι εδώ καταδικάζουμε ελπίζω να καταδικάζουμε την παράνομη ε, προσάρτηση της Κρυμαίας που έγινε πριν από δύο χρόνια. Ε, οι κατακτητές δεν κατέχουν μόνο την επικράτεια της Κρυμαίας αλλά προσπαθούν να κάνουν αυτό που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω εθνοκάθαρση ε, των Τατάρων της Κρυμαίας που είναι οι πρώτοι οι οποίοι κατηγορήθηκαν για εγκληματική δραστηριότητα. Το 1944 οι Σοβιετικοί ανακοίνωσαν ότι ε, ε, όλοι οι Τάταροι ήταν εγκληματίες και τους ε, εκτόπισαν μαζικά. Αυτό πέρασε απαρατήρητο. Από ό,τι φαίνεται η σημερινή Ρωσία προσπαθεί να επαναλάβει αυτό το έγκλημα. Οι Τάταροι της Κρυμαίας και πάλι στιγματίζονται ως εγκληματίες το βασικό τους αντιπροσωπευτικό όργανο απαγορεύτηκε και άρχισαν οι διώξεις εναντίον τους. Εμείς έχουμε εκπονήσει ένα καταπληκτικό ψήφισμα το οποίο καταγγέλει την καταστολή των ρωσικών αρχών και επίσης συνηγορεί υπέρ του συμβασμού των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ δυστυχώ να είμαι ευέλικτη αυτή τη στιγμή με το χρόνο. Θα είμαι πολύ αυστηρή. Σα ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων και τώρα ένα λεπτό ο κύριο Κοράο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Μαζική, ε, μαζικός εκτοπισμός των Τατάρων της Κρυμαίας έχει ξεκινήσει από το 1948. Πολλοί κόσμος έχει χαθεί και άλλοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στη χώρα τους παρά μόνο τη δεκαετία του 80. Οι διώξεις συνεχίστηκαν από τη Σοβιετική κυβέρνηση αλλά και από την Ουκρανική κυβέρνηση οι οποίε διαδέχτηκαν η μία την άλλη στην διοίκηση της Κρυμαίας. Ακόμα και σήμερα ε, γίνονται διώξεις ε, πολιτικών ηγετών και της μειονότητας των Τατάρων στην Κρυμαία. Αυτό που ζητάμε είναι να κλείσει αυτή η ντροπιαστική σελίδα σιωπής που έχει διαρκέσει για πολύ χρονικό διάστημα, αλλά και να κάνουμε ένα ψήφισμα στρατηγικό και πολιτικό. Είναι ντροπή που η Ευρώπη αγνοεί τις μειονότητες της Κρυμαίας, αλλά και είναι ντροπή ε, που έχει ασχοληθεί με αυτές τις μειονότητες μόνο για δικούς της στόχους. Πρόκειται για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να πάψουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Όλες οι άλλες πολιτικές σκέψεις και στρατηγικές σκέψεις θα πρέπει να περάσουν σε δεύτερο πλάνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάνοκ. Πρόεδρε, η Κρυμαία και γενικότερα η κατάσταση της κατοχής στην Ανατολική ε, Ουκρανία δεν θα πρέπει να γίνει παγωμένη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις και να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την Κρυμαία. Υπάρχουν και μειονότητες εκεί που διώκονται και ιδιαίτερα και είναι γνωστή η κατάσταση των Τατάρων, για να μην μιλήσω για τους Ουκρανούς. Ε, 20.000 έχουν φύγει και πήγαν στην υπηρετική Ουκρανία και εξωθούνται σε αποχώρηση και υπόλοιποι. Είναι μια εκδοχή του 21ου αιώνα του αναγκαστικού εκτοπισμού που έκανε ο Στάλιν το 1944. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παραμείνουν σε επαγνύπνιση και να ενθαρρύνουν την Τουρκία να υποστηρίζει τους Τατάρους ε, όπως κάνουν και με τους Τουρκομάνους στην Συρία που είναι ομοεθνείς τους όπως και οι Τάταροι ε, αυτή η πολιτική επιθετική ε, είναι απαράδεκτη ε, των 21ο αιώνα. Ευχαριστώ. Κύριε Σπαντζέρη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη φορά σε λίγους μήνες που ε, ε, μιλάμε για την υπόθεση των ε, Τάταρων και αυτό δείχνει πόσο δεσμευμένο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην, απέναντι σε αυτή τη μειονότητα που από την αρχή της κρίσης της Ουκρανίας εκδηλώσαμε την αντίθεσή μας στην προσάρτηση της Χερσονήσου από την Ρωσία. Ε, επίσης ανησυχούμε πολύ για την απόφαση που έλαβε το Δικαστήριο της Συμφερόπολης να δηλώσει ότι η Τάταρη είναι εξερμιστική οργάνωση και να τους απαγορεύσει τη δραστηριότητα. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει έντονη αντίδραση από πλευρά μας. Θα πρέπει επίσης να αναλάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμόσουμε σύντομα αυτές τις αυτό το ψήφισμα, αλλά και να αποφευθεί παρέμβαση που θα αφαιρέσει την φωνή αυτής της μειονότητας που έχει ήδη καταπιεστεί και διωχτεί πολύ στην ιστορία της. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαστάλκα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται καν να εξηγήσουμε το τι συνέβη στους ε, Ταρτάρους της ε, Κρυμαίας. Ε, δεν χρειάζεται να διευκρινίσουμε μετά του δημοψηφίσματος στην Κρυμαία, δεν χρειάζεται να εξεργήσουμε για τον εξεργασμό σε μετανάστευση, σε εκτοπισμό των Τατάρων. Σε ό,τι αφορά τις επίσημες γλώσσες στην Κρυμαία, είναι θετικά τα βήμα, είναι θετικό με πείμα αυτό, αλλά δεν ικανοποιεί όλους. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τις λύσεις αυτές ε, σε ό,τι αφορά και τις γλώσσες. Επίσης, οι πηγές ενημέρωσης δεν είναι πάντα επαρκείς και θα πρέπει να έχουμε αντίληψη το αρνητικό αντικτύπου του Ιράκ και της Ουάσιγκτον. Θα πρέπει λοιπόν να μεταβούμε εμείς εκεί και να δούμε τι γίνεται με τα ίδια μας τα μάτια. Ευχαριστώ κύριε Σπλένκοβιτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχά, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαι ικανοποιημένο με το γεγονό ότι καταλήγουμε ουσιαστικά σε μια συνένεση σε ό,τι αφορά το ψήφισμα αυτό, σε ό,τι αφορά ε, του στατάρου τη Κρυμαία, ε, μια μειονότητα τη ε, Ουκρανία που έχουν παραμείνει ε, πιστοί στην Ουκρανία μετά την προσάρτηση από πλευρά τη Ρωσία και σε ό,τι αφορά την απαγόρευση των Μέτσλης ε, της ε, Κρυμαίας το γεγονός ότι έχουν ανακηρυχθεί ε, παράνομη οργάνωση. Ε, πιστεύουμε ότι αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να γίνουν σε αυτά τα δικαιώματά τους, να απογορευτεί οποιαδήποτε είδους βίας κατά των Τατάρων της Κρυμαίας. Και θα θέλαμε στην διαδικασία επανένταξης του, τιμή, του κομματιού αυτού να ε, ακολουθηθεί η συνθήκη της Γενέβης, να επιβληθούν ε, κυρώσεις, να μετρηθούν οι κυρώσεις, ε, μάλλον εφόσον δεν έχει σημειωθεί πρόοδος και όσον δεν, είναι, δεν έχουμε εξασφαλίσει την επικράτη της Κρυμαίας. Ευχαριστώ. Κύριε Σαστραβίτσης, το 38 η Κρυμαία ήταν υποκατοχή της Ρωσίας του Τσάρου και στην πραγματικότητα προσπαθούσαν να κάνουν ένα εκρόσισμό. σεισμό. Το, το Μάιο του 1944, μετά από την του 250.000 Τατάρι, ένα ολόκληρο έθνο μεταφέρθηκε ουσιαστικά και διώχθηκε στην ε, Κεντρική Ασία. Εκατοντάδε έχασαν τον ζωή του ε, στον δρόμο ή στην εξορία. Απόλυτο λοιπόν, απόλυτη απέλαση και βλέπουμε σήμερα στην ε, Κρυμαία να συνεχίζονται αυτέ οι πολιτικοί εθνοκάθαρσεις φεύγουν από την Χερσόνησο οι Τατάροι και θεωρούνται ε, παράνομοι. Οι ακτιβίστες διώκονται, ε, καταπιέζεται ο πολιτισμός και η θρησκεία τους, κλείνουν τα μέσα ενημέρωσης και είναι σαφής ο στόχος ε, των Ρώσων. Όλα αυτά συμβαίνουν δε στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Και σε ό,τι αφορά τους ε, Μετσλής. Ε, η απαγορεύση τους γίνεται με παραβίαση διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθηθούν τα σχετικά μέτρα και τα ε, οι από πλευράς τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ήταν λάθος να μην γίνει αυτό. Δεν υπάρχει Κρυμαία, συνάδελφοι, χωρί του ταπτάρου τη Κρυμαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα περάσουμε στι πολιτικέ ομάδε. Για ένα λεπτό το λόγο για Κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να το συζητήσουμε και το συζητάμε σήμερα για δεύτερη φορά. Από το Φεβρουάριο έχει επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση των Τατάρων. Ε, ε, το σώμα τους ε, απαγορεύθηκε το αντιπροσωπευτικό το ΜΑΙΛΙΣ, το χαρακτηρίστηκαν εγκληματική οργάνωση η Κρυμαία είναι ε, έδαφος της ε, Ουκρανίας που παράνομα προσήρτησε η Ρωσία. Η Τάταρη είναι ε, μια πάρα πολύ ενεργή και δραστήρια κοινότητα. Εμεί δεν αναγνωρίζουμε την προσάρτηση αυτή. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ε, και να αρχίσουν και διαπραγματεύσεις που να αναγκάσουν τη Ρωσία να αποχωρήσει. Οι ε, διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην Κρυμαία για να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ 1,5 λεπτό κύριο Χάουιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απόφαση να ανασταλεί η λειτουργία του Μέισλης στην Κρυμαία είναι κατάφορη παραβίαση του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε. Ε, κρατούνται οι τάταροι, ε, τους παίρνουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα και το DNA. Είναι νέα ο κύμα αυτό ε, παραβίασης των δικαιωμάτων και δίωξης ε, των τατάρων. Τους εκτόπισαν ε, σε μακρινές περιοχές της Σοβιετικής τότε Ένωσης ε, θα πρέπει ε, διπλωματικά να κάνουμε διαβήματα προς τη Ρωσία ε, για να σεβαστεί ε, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και την αντίστοιχη σύμβαση του ΟΗΕ. Συναντήθηκα στο Κίεβο με ένα από τους δύο ηγέτες που διώκονται. Τους είπαμε ότι δεν θα τους ξεχάσουμε και θα υπεθυμίσουμε σε όλη την Ευρώπη τα δεινά που υφίσταται. Ένα λεπτό, ο κύριος Δημέσμακερ. Τι είναι το σπίτι, συνάδελφοι. Είναι ο ορισμός των Αμερικανού συγγραφέα Κλαρίς Εμχάν. Το σπίτι είναι ένα ασφαλές μέρος όπου δεν φοβάται κανείς για επιθέσεις, για ασφαλείς σχέσεις και επιβεβαίωση. Δυστυχώ όμως για τους ατάρσεις της Κρυμαίας η πατρίδα τους, το σπίτι τους δεν είναι πλέον αυτή η ασφάλεια. Έχουν ζήσει απελάσεις, γενοκτονίες, ένα από τα πια βία καθεστώτα του 20ου αιώνα με συνεχή καταπίεση των δικαιωμάτων τους και κανεί δεν περίμενε ότι τον 21ο αιώνα ένα κράτο, ένα μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ με τέτοιο κατάφορο τρόπο θα παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα και σήμερα οι Ταρτάροι της Κρυμαίας είναι εκ νέου θύματα αυτού του καθεστώς. Ε, απαγωγές, στράτευση καταναγκαστική στο ρωσικό στρατό, καταπάτηση των δημοκρατικών αξιών τους. 20.000 από την Κρυμαία, 5.000 από τη Σεβαστόπολη αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν. Και στην, ε, στο ψήφισμα τονίζουμε την ευθύνη του Κρεμλίνου, αλλά ζητάμε να μην σταματήσει η πίεση και σε εμά να διατηρήσουμε τις ε, κυρώσει, γιατί υπολογίζουν σε εμά αυτό ο περήφανο λαό. Ευχαριστώ, κυρία Σχάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Η παράνομη προσπάθηση τη Κρυμαία από του Ρωσού οδήγησε στην καταπάτηση των δικαιωμάτων και κάποιων μειονοτήτων όπω η Θαθάρη οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν και ως τρομοκράτες, αντιμετωπίζουν βία, απαγωγές, δολοφονίες και οι απονομαζόμενες αρχές δεν διώκουν τους υπευθύνου. Το, η οργάνωση, το σώμα του μέλησε πλέον απαγορεύεται και εξαναγκάζονται σε εξορία. Οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στον ΟΑΣΑ, στον ΟΗΕ, στα δικαιώματά τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αποτελούν ε, άλλο ένα κακό σημάδι και η καταπολέμηση, η απαγόρευση της ελευθερίας έκφρασης. Όλα αυτά λοιπόν κατά πίεση των ε, Τατάρων της Κρυμαίας θα πρέπει να λάβει ένα τέρμα, όπως και η παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας συνολικά. Ευχαριστώ. Κύριε Σαφχάουζερ, για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά ε, συνένεση στο σφάλμα. Οι Τάταροι είναι εθνότητα ε, στην Κρυμαία. Ε, ε, το υποτιθέμενο καθεστώ αυτοκτόνων λαών θα τους έδινε περισσότερα δικαιώματα. Μπορεί να διώχθηκαν από το Στάλιν, αλλά όλος ο Ουκρανικός λαός, όλοι οι λαοί, η Μάιζελη λέει, που είναι η κοινοβουλευτική του συνέλευση Ισλαμική, λέει ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους Ρώσους, Γερμανού Έλληνε, Αρμενίου στην Κρυμαία, ε, λόγω μιας ιστορικής αμφισβητήσιμης παρουσίας, γιατί πρώτοι βρέθηκαν σε αυτή τη χερσόνηση. Το Μάιλις ποτέ δεν αναγνωρίστηκε από καμία Ουκρανική αρχή πριν ε, ε, ενωθεί ε, με την Ρωσία. Ο Γκολοβάτη, υπουργό τη 14 Μαρτίου του 1987, απαντώντα στο Κοινοβούλιο, είπε ότι είναι παράνομη η δράση Μάιλις στην Ουκρανία. Έγινε εγκληματική τρομοκρατική οργάνωση και στο Κέρσοφ έχει ε, ε τους γκρίζους λύκους και άλλες τέτοιες τουρκικές οργανώσεις. Ε, ένα λεπτό, ο κύριος Κόρβεν Μίκε. Ευχαριστώ. Πήγα στην Κρυμαία και μίλησα με εκπροσώπους των Τατάρων εκεί και με, με απλούς ανθρώπους στο δρόμο. Οι Τάταροι ήταν υπέρ των Ρώσων και ε, ήταν πάρα πολύ απογοητευμένοι ε, γιατί θεωρούσαν ότι η κατάστασή τους θα βελτιωνότανε, η οποία όμως δυστυχώς επιδεινώθηκε. Στην Ουκρανία είναι οι ίδιοι που παραμένουν στην εξουσία και οι ίδιοι που εκμεταλλεύονται εκεί και λιμένονται την κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα και με τους Τατάρους στην Κρυμαία ε, ε, η βουλή τους στο Μέιλις θεωρείται εγκληματική οργάνωση και είδαμε τι έγινε και το χειμώνα. Είχε κοπεί το ρεύμα στην Κρυμαία ε, και η βουλή των Τατάρων ήταν υπέρ της κατάστασης αυτή. Λοιπόν, τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα, δεν είναι καθόλου απλά. Και κατά τα άλλα, όπως ξέρετε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαλυθεί. Ο κύριος Στέτινα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, τον Μάιο του 1944 ο Στάλιν εξόρισε 350.000 Τατάρους στο Ουσμπεκιστάν. Πάνω από 10.000 έχαναν τη ζωή τους από αυτήν την υποχρεωτική καταναγκαστική μεταφορά. Οι πολίτες λοιπόν ταταρικής καταγωγής στην Κρυμαία δυστυχώς είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και οι ρωσικές αρχές κατοχής τους θεωρούν ακριβώς κατώτερους και θέλουν να τους διώξουν από την Κρυμαία. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε την τραγωδία του σταλινικής περίοδου. Την επόμενη εβδομάδα εγώ θα πάρω μέρος σε μια εκδήλωση στο Κίεβο ε, για την γενοκτονία των Τατάρων και θα καταθέσω στον κύριο Τσουμπάρ, τον πρόεδρο της Μαζλής, ε, ε, το ψήφισμά μας. Η κυρία Φώτιγκα. Η αλήθεια είναι ότι η Κρυμαία είναι θα έλεγα το σημείο από τα οποία όλα ξεκίνησαν για τους Τατάρους πάντα ήσαν πολέμοι της βαρβαρότητας των Ρώσων οι Τάταροι. Πάντα πολέμησαν και τον Στάλιν και ακόμα και σήμερα η Κρυμαία μετά από την προσάρτησή της στη βίαιη από την Ρωσία δημιουργεί προβλήματα στους Τατάρους. Το ίδιο ίσως να συμβαίνει και για άλλες μειονότητες, αλλά το εύρος της βαρβαρότητας των Ρώσων εις βάρος των Τατάρων είναι κάτι το απαράδεκτο. Ο Χατζημιλεύ ο υπεύθυνο ε, εκπρόσωπός τους, ε, θεωρεί ότι εξακολουθεί η κατηγορία αυτή των πολιτών να είναι θύμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να σταματήσει η παράνομη προσάρτηση ε, της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Θα πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία και μέχρι να γίνει αυτό υποχρεούται να προστατεύει το λαό της Κρυμαίας η Ρωσία από οποιαδήποτε διάκριση και ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, Δυστυχώ το αντίθετο παρατηρούμε. Η απαγόρευση της Μαϊλής και η δίωξη των μελών της είναι πραγματικά λυπηρή και θα πρέπει να τερματιστεί. Σύντομα, ε, προσεχώ θα συζητήσουμε πάλι του υποψηφίου για το βραβείο Ζαχάροφ. Βλέποντα την κατάσταση των Τατάρων στην Κρυμαία, θα πρότεινα να σκεφτούμε ε, έναν από του υποψηφίου, τον Μουσταφά Τζεμίλευ, που είναι ηγέτη των Τατάρων τη Κρυμαία και του έχουν ε, απαγορεύσει την είσοδο λόγω δραστηριοτήτων που είχε στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τατάρων στην Κρυμαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν ε, ανεχόμαστε την παρούσα προσάρτηση ε, της Κρυμαία και την καταστολή των Τατάρων της Κρυμαία. Ευχαριστώ κύριε Σόγκορ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ θα μιλήσω ουγγρικά. Η, η η συνέλευση των Κρυμαίων Τατάρων καταδεικνύει το πώς λειτουργεί η ρωσική πολιτική. Με τον νόμο κατά του εξτρεμισμού αποφάσισε η Ρωσία να κλείσει αυτή τη λαϊκή συνέλευση και έκανε όλη την ε, μειονότητα των Τατάρων κατά την άποψή τους εξτρεμιστές και επικίνδυνους για την Ευρώπη. Όλα αυτά γίνεται, γίνονται μέσα στην προσπάθεια των ε, Ρώσων να διεκδικήσουν δικαιώματα αυτονομίας για τους Ρώσους που βρίσκονται στην Ανατολική ε, Ουκρανία. Αυτό που κάνουν με τους Τατάρους Κρυμαίας το δείχνουν πόσο χωρί νόημα είναι αυτή η διεκδίκηση των Ρώσων για την Ουκρανία. Εμεί δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα κράτο μέλο να εφαρμόσει το ίδιο τέχνασμα για να θεωρήσει συλλογικά μια ολόκληρη κοινότητα εξτρεμιστέ. Δυστυχώ οι Ρώσοι έχουν κάνει προσπάθειε προ την κατεύθυνση αυτή. Δεν μπορούν οι ηθαγενεί ομάδε να θεωρούνται ξένο σώμα. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα το οποίο δημιουργεί τεράστιε κοινωνικέ εντάσει. Ευχαριστώ πολύ ακολουθεί η προσάρτηση της Κρυμαίας από τους Ρώσους το 2014 και η, ο χαρακτηρισμός τους ως, τρομοκράτε ως τρομοκράτες έχει οδηγήσει σε μεγάλα βάσανα στην κοινότητα των Κρυμαίων Τατάρων. Πολλοί από αυτούς είναι στη φυλακή, άλλοι έχουν βασανιστεί. Είναι η μόνη μειονότητα στην Κρυμαία που είναι αυτόχθον και η οποία με έναν τρόπο ο οποίος είναι οργανωμένος αντιστέκεται στη ρωσική ε, ομοσπονδία και δεν θέλει τη ρωσική κατοχή. Κάνω λοιπόν μια πρόσκληση, μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κάτι μέλη της να παγώσουν τα στοιχεία ενεργητικού αυτών που έχουν συμβάλει στην προσάρτηση της ε, ε και να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να ε, απελευθερώσουμε τον πληθυσμό της περιοχής αυτής. Η ενέργεια αυτή έτσι κι αλλιώς απειλεί και την ασφάλεια της Ευρώπης γιατί έχει στρατικοποιηθεί οι χερσόνες που έχουν εγκαταστήσει σύγχρονα α, οπλικά συστήματα και αυτό είναι απειλή για την Ευρώπη. Ζητώ συγγνώμη. Σα είπα ότι έχουμε πρόβλημα χρόνου. Μόνο δύο μιλητέ βάσει τη διαδικασία Catch και λυπάμαι για αυτού οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν. Ο χρόνο ρέει εναντίον μα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μια έκθεση η οποία περιγράφει νομίζω καλά την κατάσταση στην Κρυμαία μετά την προσάρτηση ε, της περιοχής από την Ρωσική Ομοσπονδία. Υπάρχει συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά και η απαγόρευση λειτουργίας της Μαζλής είναι κάτι το απαράδεκτο ε, και κατηγορούνται τώρα τα μέλη του Μαζλής για ακραίο εξτρεμισμό και ε, για σαμποτάζ της χώρας, υπονόμευση της χώρας. Δεν διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε από πάρα πολύ κοντά την κατάσταση, ιδιαίτερα σχετικά με τα ΜΚΟ, γιατί εγώ συναντήθηκα με σημοσιογράφους οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την περιοχή αυτή και γι' αυτό ακριβώς είμαι υπέρ πέμπτη έκθεση αυτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για τους Τατάρους της Κρυμαίας και την ε, κατάρριξη της ε, Μαϊτζλής καταδεικνύει την ε, βία και την διάκριση που ασκείται εναντίον τους. Υπάρχουν κατασταλτικά μέτρα από την Ρωσική Ομοσπονδία. Τους απαγορεύεται να ταξιδέψουν πέρα από την περιοχή τους. Δεν υπάρχει πλέον δικαιοσύνη. Έχουν χαρακτηριστεί εξτρεμιστές και οι ηγέτες της κοινότητας των Τατάρων είναι στη φυλακή η υποδίωξη. Δεν τους επιτρέπεται σε αυτούς που είναι εκτός της χερσονήσου Κρυμαίας να εισέλθουν εκεί. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αντιδράσει, αλλιώς θα μείνουμε απλώς παθητικοί θεατές μιας παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. Πρέπει να σταματήσει η καταστολή στη χερσότσο της Κρινέας και η παραβίαση των απαράγραπτων δικαιωμάτων. Έχει κλείσει ο κατάλογος και δίνω το λόγο στην Επίτροπο την κυρία Γιούροβα να απαντήσει. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο χρόνια μετά από την παράνομη ένταξη της Κρυμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε τις βαθύτατες ανησυχίες της για την ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Χευσόνησο της Κρυμαίας. Στέρηση ελευθερίας έκφρασης, επίσης ελλείψεις στον τομέα του σεβασμού των θρησκευτικών δικαιωμάτων, των μειονοτικών δικαιωμάτων και φυσικά μέτρα εις βάρος των Τατάρων της Κρυμαίας. Η κυρία Μογκερίνη τα συζήτησε, τα έθεσε τα θέματα αυτά και συναντήθηκε με εκπροσώπους των Τατάρων της Κρυμαίας στην επίσκεψή της στο Κίεβο τον Νοέμβριο του 2015 η απόφαση της 26ης Απριλίου για την απαγόρευση της λειτουργίας του Μαϊσλής, το οποίο είναι ε, το σώμα που εκπροσωπεί τους Τατάρους, είναι μια επίθεση βίαιης βάρος των δικαιωμάτων των Τατάρων στο σύνολό τους. Είναι ε, μια επιπλέον λοιπόν σημαντική χειροτέρευση της κατάστασης στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Χερσόνησο ε, της Κρυμαίας μετά από την παράνομη προσάρτησή της από τη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014. Να επαναλάβω λοιπόν για μια ακόμη φορά την ξεκάθαρη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ανεμπόδιστη ε, πρόσβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εξετάζουν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή της Κρυμαίας και της Σεβαστούπολης. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, στις 18 Μαΐου, ε, θα υπάρξουν ε, τελετές για τον εκτοπισμό των Τατάρων το 1944. Πέρυσι δεν μπόρεσαν να οργανώσουν ειρηνικέ εκδηλώσεις οι Τάταροι για, το ίδιο θέμα. Νομίζω ότι αυτό μας υπενθυμίζει ότι οι κάτοικοι αυτοί της Κρυμαίας έχουν υποφέρει ιστορικά και οι διώξεις εις βάρος τους θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Σας ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ τους συναδέλφους, έχω επτά